Bene, cominciamo subito i nostri lavori anche perché abbiamo pur avendo un'ora e mezza a nostra disposizione, il dibattito però... Η συζήτηση έχει σημασία βέβαια και θα ήθελα να ξεκινήσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, ευχαριστώ και τον κύριο Σίμψον όπως επίσης και τους εκπροσώπους της Επιτροπής ΣΥΤΡΑ για αυτή την τέταρτη μεικτή συνάντηση ανάμεσα στην Επιτροπή μας και την Επιτροπή Μεταφορών. Μια συνάντηση που θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε κοινά θέματα. Η συνεδρίαση αυτή όπως γνωρίζετε επί τη βάση του κανονισμού προεδρεύεται και από τους δύο προέδρους, συμπροεδρεύεται δηλαδή, αλλά για να διευκολυνθούν οι εργασίες θα προεδρεύσω εγώ, πάντα όμως μαζί μου με τον κύριο Σίμψον που θα παίρνει το λόγο όποτε το επιθυμεί. Γνωρίζετε ότι έχουμε 753 τροπολογίες. 753 τροπολογίες που έχουν ήδη κατατεθεί θα μας παρουσιάσουν επίσης και τα τρία προηγούμενα πρακτικά των συνεδριάσεών μας και θα ακολουθήσει η συζήτηση. 27 Νοεμβρίου προβλέπεται η αποκοινού ψηφοφορία. Και θα ξεκινήσω αμέσως τις εργασίες μας. Για πέντε λεπτά θα δώσω το λόγο στην πρώτη συγγήτρια, την κυρία Γιάλα Σεντέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να πω ότι χαίρομαι τελικά που βρίσκομαι εδώ, που βρισκόμαστε όλοι εδώ όλες τις δυσκολίες. Είναι περίπλοκο βέβαια να κανονίζουμε κοινέ συνεδριάσεις. Ε, μας ε, ζητήθηκε ευελιξία αυτή τη φορά. Ε, προσπαθήσαμε και πράγματι δεχτήκαμε να αναβάλουμε για την ε, τρίτη το θέμα του συνδέοντας την Ευρώπη έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ε, παρουσία. Ελπίζω στο μέλλον η γραμματεία θα δείχνει μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε ε, να διευκολύνει στα, την εργασία μας. Κάθε φορά που ζητούμε αλλαγές μας τις αρνούνται. Ε, η πολιτική όμως είμαστε εμείς και ελπίζω την επόμενη φορά η Γραμματεία να κάνει μια, καλύτερη, μια μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι ώστε να μας ε, διευκολύνει. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο η ψηφοφορία να γίνει την Τρίτη να είναι παρόντες πιο πολύ βουλευτέ. Τώρα, σε σχέση με τον μηχανισμό, με τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, ε, έχουμε ανταλλάξει απόψεις και η Κυπριακή Προεδρία είχε υποβάλει έναν προϋπολογισμό πραγματικά καθόλου ικανοποιητικό γιατί μετά τις αποφάσεις και τις ε, γενικές δηλώσεις υπέρ της ανάπτυξης ε, και της ε, απασχόλησης στην Ευρώπη, δεδομένης και της κατάστασης κρίσης, ανεργίας κλπ. που επικρατεί, ε, η Κυπριακή Προεδρία ε, που η για πρώτη φορά προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έδωσε αρκετή σημασία οικονομικά εννοώ, χρηματικά σε αυτό το κείμενο το οποίο είναι μοχλός πραγματικά και θα έλεγα ε, ταπεινό σχετικά ε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό που χρειάζεται. Παρόλα αυτά ε, η Κυπριακή Προεδρία μας παρουσίασε ένα προπολογισμό ανεπαρκή, δεν το δεχόμαστε. Απορρίπτουμε αυτή την πρόταση της Προεδρίας περί μεγάλης περικοπής του προπολογισμού της διευκόλυνσης αυτής οι εισηγητέ είχαμε συμφωνήσει ε, αν το Συμβούλιο περικόψει μεγάλο ε, ποσοστό ε, είχαμε συμφωνήσει να ξαναδούμε τον κατάλογο των σχεδίων, των project. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πολεμήσουμε για να διατηρήσουμε τον προπολογισμό μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, Έχουμε κάποιες ακραίες ε, προτάσεις περί ριζικής αναδιάρθρωσης του κειμένου, δεδομένου και του αυτού που μόλις είπα κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Υπάρχουν όμως άλλες τροπολογίες που ε, επιδιώκουν να ε, αυξηθεί κατά 5% η χρηματοδότηση του συνολικού δικτύου. Ε, Παρ' όλα αυτά, η, ε, ο προπολογισμό είναι περιορισμένος ε, και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το ε, πετύχουμε. Μετά υπάρχουν κάποιες Ιρλανδικές τροπολογίες για την ειδική περίπτωση της Ιρλανδίας που είναι νησί και για τις συνδρομικές μεταφορές προβλέπουν τη δυνατότητα σε ορισμένα κράτη-μέλη, αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, να ε, δεχτούμε τη χρηματοδότηση και αυτών των δικτύων. Αυτό μπορούμε να το ε, συζητήσουμε, παρόλο ότι έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης. Ε, σε ό,τι αφορά τα αστικά, τους αστικούς κόμπους, είναι επίσης πολύ σημαντικό που, ετέθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που μας υποστήριξαν. Σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, καταλαβαίνω ε, ότι κάποιοι συνάλφοι ε, θέλουν να χρηματοδοτηθούν κάποιες τεχνολογικές ε, πτυχές που έχουν πιο πολύ σχέση με τον ορίζοντα 2020, 2020. Και για κάποια πολύ συγκεκριμένα σχέδια ε, με συνέργειες μεταξύ των τριών τομέων. Ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και να δεχτούμε τις προτάσεις, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες, περιοχές, ε, ε, πολύ συγκεκριμένες ε, ε, περιπτώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης ε, του τροχαίου υλικού, προτάσεις από τη Γερμανία. Ο προπολογισμό είναι πολύ περιορισμένος, σας το έχω πει. Ε, αναφέρεται ο αποκανονισμός πιο πολύ βασικά στις υποδομές, οπότε ε, θα ε, ήθελα να χρησιμοποιηθούν ε, χρηματοδοτικά μέσα, χρηματοοικονομικά μέσα και όχι η χρηματοδότηση από αυτόν τον κανονισμό. Ε, τέλος, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης, Ε, με κάποιες ελάχιστες εξαιρεσει, όπως για παράδειγμα οι θάλασσε λεωφόροι που θα μπορούσαμε να δεχτούμε μια αύξηση ε, και για την ε, συνοχή έχουμε κάνει μια συμβαστική πρόταση που νομίζω κινείται προς σωστή κατεύθυνση προς την κατεύθυνση της Περιφερειακής Επιτροπής και των συναδέλφων από τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε Καταρχήν, να διατηρήσουμε την εθνική κατανομή, καταρχήν λέω, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλουν προγράμματα όλες οι χώρες και μετά όταν εντοπιστούν οι κίνδυνοι και έχουμε και την τεχνική συνδρομή να περάσουμε στην ε, επιλογή των πιο σημαντικών σχεδίων, των πιο αποδοτικών, ε, των πιο ανταγωνιστικών σχεδίων. Ε, τέλος, συνέργεια. Συνέργεια είναι πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν βέβαια είναι διστακτική πολλές φορές, αλλά Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, έχουμε μια, ένα κανονισμό με περιορισμένο προπολογισμό και γι' αυτό το λόγο ειδικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ τομέων που συνδέονται μεταξύ του τόσο πολύ τηλεπικοινωνίας, μεταφορές, ενέργεια. Ευχαριστώ. Ο Ρικέ το λόγο. Παρακαλώ σεβαστεί το χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Λέει ο κύριος Ρικέ, δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν ήδη. Νομίζω ότι όλοι και οι συγητές και οι βουλευτές που κατέθεσαν τροπολογίες επιδιώκουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τον στόχο της ανάπτυξης. Αυτό το μέσο είναι το καλύτερο που έχουμε για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ας μείνουμε πιστοί λοιπόν σε αυτό το στόχο και ας επιδιώξουμε την ανάπτυξη σεβόμενη το περιβάλλον με ταχύτητα και επίσης τα διαφορετικά ταμεία. Μία πρόταση τώρα, για, μια, ένα σχόλιο μάλλον για την κυπριακή πρόταση. Η συνάδελφος ε, θα μας πει αν είναι ικανοποιημένη στα θέματα της ενέργειας. 22,5 δις, από τα οποία 7,5 συνοχή, 15 δις για νέες προτάσεις. Αυτό είναι μηδενική πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν. Στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο είχαμε 10 δις. Αν επικαιροποιήσουμε τα ποσά αυτά και τα ενημερώσουμε, τότε η πρόταση που κάνει η Κυπριακή Προεδρία είναι μηδενική. Όχι απλώς δεν γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη, αλλά ακυρώνονται οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει. Η πρόταση αυτή δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεν συνιστά καν βάση για συζήτηση. Ας περάσω σε κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα. <clears throat> Το πρόβλημα του Ταμείου Συνοχής το ανέφερε και η Ινές. Έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία σέβεται τις εθνικές προτάσεις, δέχεται επίσης πάντα τη συνέχιση της διαδικασίας κεντρικού ελέγχου, τώρα για να ευνοήσουμε ορισμένους τρόπους αηφόρου ε, μεταφορών, αηφόρων μορφών μεταφορών όπως οι θαλάσσιες λεωφόροι, οι σιδηρόδρομοι κτλ. Η διευκόλυνση της αμοιβαίας πληροφόρησης και ενημέρωσης όπως επίσης και η συνεργασία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα γιατί χάνουμε πάρα πολύ ενέργεια σε ε, μορφές επιτροπολογίας και να διατηρήσουμε επίσης ανοιχτό και το επίπεδο περιφερειακής διαβούλευσης μέσω απλούστευσης των διαδικασιών να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο να μην είναι πάρα πολύ ε, βαρύ θα έλεγα να καθορίζει με συγκεκριμένο τρόπο κάποιες ποσοστώσεις ε, οι οποίες ε, να έχουν σημασία και βάρος και αυτά όλα βρίσκονται στις προτάσεις των ποσοστών που κάνουμε εμείς και να μην μείνουμε στο επίπεδο του συμβολικού και του ασήμαντου. Γι' αυτό που θα ονόμαζα έκυπνο ε, ομπαρκέ, ε, σαν παράδειγμα καταμέτρηση ε, θορύβων, ασφάλεια, μέτρα ασφαλείας κτλ. Ό,τι δηλαδή βρίσκεται σε, σε οχήματα, σε σκάφη, σε αεροσκάφη αλλά δεν είναι ε, αποκλειστικά τμήμα αυτών των ε, υποδομών. Είναι κάτι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο ε, ποσό. Βέβαια στο σύνολο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα ποσά είναι σημαντικά και απευθύνεται σε εξωθεσμικούς θα έλεγα στην εξωθεσμική λεγόμενη ζήτηση δεν εντάσσεται στην περίμετρο των δικών μας προβλέψεων. Για τον θόρυβο έχει τεθεί το θέμα, υπάρχουν χώρες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό να κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε ότι το ενδιαφέρον ποικίλει πάντως από χώρα σε χώρα. Υπάρχει διαφοροποίηση επίσης και σε επίπεδο ζήτησης για σιωδρομικές εμπορικές μεταφορές και θα πρέπει να βρεθούν άλλου είδους λύσεις από αυτές τις οποίες έχουμε μέχρι τώρα καταλήξει. Εδώ οι συζητήσεις συνεχίζονται. Στα παραρτήματα θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη για τον σεβασμό των κριτηρίων. Θα πρέπει επίσης να παραμείνουμε στην ουσία, πάντα στοχεύοντας με τα δίκτυα αυτά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Να είμαστε φυσικά πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την, με τον όρο <clears throat> αποτελεσματικότητα και κόστος, γιατί δεν έχουμε πολλά χρήματα. Και ε, να ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν ε, και άλλες μορφές χρηματοδότησης τις οποίες θα πρέπει να ανοιχνεύσουμε. Εφόσον παραμείνουμε λοιπόν στα πλαίσια αυτά, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε γιατί παρά τις διαφορές υπάρχει φυσικά, υπάρχει φυσικά επιθυμία για συμφωνία και ο βασικός ένοχος φυσικά είναι το Συμβούλιο. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Η κυρία Βάλε αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σχεδεσηγητές και τους βουλευτές οι οποίοι βοήθησαν να βελτιωθεί η έκθεση. Ελλάδα με γύρω στη, σχεδόν στις 600 ε, τροπολογίες ε, και βεβαίως ε, αναμένω και τους γεωδησηγητές για να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Από την σκοπιά της Επιτροπής Βιομηχανίας χαίρομαι για το ότι οι περισσότεροι στηρίζουν την ε, άποψη της εισηγητού για την χρηματοδότηση των τομέων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Όσον αφορά τώρα την πρόταση τη Κυπριακή Προεδρία, είναι απαράδεκτη, συμφωνώ με του συναδέλφου, και σημαίνει περικοπή κατά 40%. Ξέρω πω οι πόροι βεβαίω ε, σπανίζουν ε, αυτή την εποχή, αλλά το μήνυμα που στέλνουμε στου πολίτε και στι αγορέ πρέπει να είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι ε, μια συνεχής λιτότητα και να μην βεβαίω αντιβαίνει και τη νέα κατεύθυνση που έθεσαν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι πολίτες για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να βγούμε από την ύφεση. Επίσης, μαζί με τους συναδέλφους μου υποστηρίζω την αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν για 50 δισεκατομμύρια ευρώ και είμαστε πεπισμένοι για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του κάθε ευρώ αν θέλουμε να εξορνήσουμε τις υποδομές μας. Και θεωρώ πως ε, την θέση μας θα την στηρίξουν και οι συνάδελφοι ε, από όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, μεταφορών, βιομηχανίας, προϋπολογισμού. Βεβαίως έχουμε ευθύνη για να διασφαλίσουμε την πιο αποτελεσματική χρήση του μέσου αυτού. Με τους περιορισμένους πόρους βεβαίως χρειάζεται, χρειάζονται εργαλεία μόχλευσης για να έχουμε και ιδιωτική χρηματοδότηση, οπότε δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις δημόσιες επιδοτήσεις. Γι' αυτό ο τομέας της ενέργειας είναι αυτό στον οποίο συνιστούμε 80% του προπολογισμού να πάει σε έργα κοινή ωφελία μέσω τέτοιων χρηματοδοτικών μέσων. Και χαιρόμαστε για το ότι οι κύριοι Πυρίλιο Τέρμς, Κάντσιαν και λοιποί ε, έχουν καταθέσει ποσοστά μεταξύ 90 60 και 90% και είμαι σίγουρο πως θα βρεθεί μια συμβαστική λύση. Όσον αφορά τις λεπικοινωνίες θεωρούμε πως το βάρος πρέπει να δοθεί στο να δημιουργήσουμε ζήτηση για την ευρυζωνικότητα, κάτι το οποίο στηρίζει και η κυρία Τροτμάν και ο κύριος Πυρίλιο Μετροπολογίες τους και ο κύριος Κάντσιαν κατέθεσε τροπολογίες για να πάει να, η χρηματοδότηση να προσανατολιστεί προς τα μέσα αυτά, όμως εκφράσαμε την άποψη πως η πλειοψηφία της χρηματοδότησης των υποδομών αυτών, όπως της Ευρωπαϊα, Οριζοντίων Προτεραιοτήτων κτλ., πρέπει να γίνει μέσω επιδοτήσεων για το άρθρο 10, για τα ποσοστά χρηματοδότηση. Είχαμε πολλές τροπολογίες από του συναδέλφους Ε, ποσοστά χρηματοδότησης ε, μεταξύ 50 και 80% και νομίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες ε, για το ποσοστό της συγχρηματοδότησης. Να σας μεθυμίσω εδώ πέρα πως στόχος σε αυτούς τους δύο τομείς είναι να διασφαλίσουμε πως η αγορά θα παραμείνει στο κέντρο της διαδικασίας, να μην έχουμε στρεβλώσεις και κεντρικές ε, πολιτικές αποφάσεις. Επίσης, να υπενθυμίσω εδώ πέρα πως δεν έχουμε άλλη μια εκδοχή των διαρθρωτικών κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Είχε σχεδιαστεί ω ένα αναπτυξιακό μέσο άλλης φύσης που θα μπορούσε να συμπληρώνει την παραδοσιακή χρηματοδότηση. Αυτή ακριβώς είναι η ε, αλλαγή νοοτροπίας ε, η οποία απαιτείται και από εμά βεβαίω εάν είναι να λειτουργήσει. Τις ερχόμενε εβδομάδε. θα πρέπει να αγωνιστούμε για τον προπολογισμό, αλλά πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι και να αναδιατάξουμε τις προτεραιότητες μας σύμφωνα με τα μέσα που έχουμε. Αν οι ευρωπαϊκοί πόροι περικοπούν, θα πρέπει να έχουμε πολιτικές επιλογές για το τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Αλλιώς δεν θα έχουν και κανένα αντίκτυπο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες μας, είτε ολοκλήρωση της αγοράς, είτε ασφάλεια, ενεργειακή, είτε ενσωμάτωση των ΑΠΕ, είτε να διαλέξουμε μία προτεραιότητα ανά Όσον αφορά δε, τα κριτήρια ανάθεσης προτείνονται στο άρθρο 17, νομίζω μπορούμε να στον και με τα πολυετή προγράμματα εργασίας κομισιών. Οι επιλογή λοιπόν είναι σκληρέ, συνάδελφοι, αν είναι η ευθύνη μας ως Κοινοβούλιο να ορίσουμε πολιτικές προτεραιότητες και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερο τρόπο του διαθέσιμου πόρου. Και βεβαίω αναμένουμε γωνία τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φέρν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να αναφέρω την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας. Πολλοί συναδελφοί είπαν κάτι ε, σχετικό. Δεν θα σταθώ πολύ. Να πω ότι όσο περισσότερο κόβουμε τον προϋπολογισμό τόσο πιο δύσκολο θα είναι να έχουμε έναν καλό προϋπολογισμό. Γιατί όλοι ε, μένουν σε αυτά τα οποία ήδη έχουν, είτε μιλάμε γεωργία, ταμεία συνοχής κτλ. Αλλά ποιος θα υπερασπιστεί πραγματικά τις δαπάνες που χρειάζονται για να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία για το μέλλον, καινοτομία, υποδομέ κτλ. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Για τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Περιπολογισμού για το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη, κάποια σχόλια κυρίω για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Είναι θετικό κατά την άποψη τη Επιτροπής μα πω ε, τα μέσα αυτά έχουν γίνει δεκτά από την εισηγήτρια η όλη η σύλληψή τους. Κάποια τεχνικά σχόλια. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε την λέξη για τις επενδύσεις ε, ε, λιγότερο από βελτιστές κάτι το, και σε ορισμένα σημεία το sub έχει μείνει non-optimal, το οποίο ακούγεται βεβαίως πολύ αρνητικότερο, δεν πρέπει να τρομάζουμε τους επενδυτές. Το ίδιο ισχύει και για τη στρέβλωση της αγοράς δεν θέλουμε εδώ πέρα πραγματικά να αφήσουμε έξω άλλες μορφές κρηματοδότησης. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά θέλουμε εδώ πέρα να υπάρξει μία αγορά για επενδυτές οι οποίοι δεν επενδύουν οπωσδήποτε σε αυτά τα προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλάμε δηλαδή πάρα πολύ για στρεβλώσεις. Να σκεφτούμε λίγο και το, το μέλλον, τη σημασία της συμπληρωματικότητας κτλ. Και εδώ πέρα νομίζω έχουμε κάποιες καλές τροπολογίες από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Επίσης θα ήθελα να τονίσω λίγο το εξής η έκθεση πρέπει να σταθεί λίγο στον στόχο που έχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Το πρόβλημα με την οικονομική μας κατάσταση είναι το εξής. Πολλές καλές επενδύσεις δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε πίστοση, περιορισμοί, υπάρχουν στράψες κτλ. Και έτσι δεν υπάρχει οικονομική ανάκαμψη. Για εμάς η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ένα υψηλό ποσοστό μόχλευσης είναι ουσιαστική σημασίας και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο προσωρινό μέτρο, αλλά θα ε, το χρειαστούμε και μακροπρόθεσμα. Νομίζω πρέπει να το τονίσουμε αυτό λίγο παραπάνω. Επίσης, θεωρούν πω είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αξιολογείται το μέσο αυτό η Κομισιόν να προτείνει μελλοντικά βήματα. Τι θα κάνουμε δηλαδή για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι επενδύσεις σε έργα προτεραιότητας. Εμείς προτείναμε παραδείγματο χάρη να δούμε την ιδέα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, επενδύσεις σε ΑΠΕ κτλ. Μπορούμε επίσης να απτύξουμε διάφορα μέσα μετοχικού κεφαλαίου. Ε, πάρα πολλά υπάρχουν στη διάθεσή μας για τις μελλοντικέ αυτές προοπτικές. Επίσης δείτε και την πρωτοβουλία των ομολόγων έργου που τονίσαμε σε κάποιες προτεραιότητες μας το θέμα δε αυτό της ανάμιξης επιχορήγησης με ε, χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρέπει να έχουμε κάποια εργαλεία στη διάθεσή μας, κάποια έργα μπορεί να χρησιμοποιήσουν τυχή στήριξη, κάποια άλλα, κάποια άλλη, κάποιο άλλο είδους χρηματοδότηση. Ας έχουμε λοιπόν, να ανοιχτή στέση όσον αφορά την μεικτή χρηματοδότηση. Τέλος για τη συνοχή. Το αναφέραμε, είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε την συμπερίληψη της χρηματοδότησης της συνοχής στο μέσο αυτό, γιατί η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία υπάρχει όχι μόνο για τις πλουσιότερες δυτικές χώρες, αλλά και για τις χώρες της συνοχής. Αλλά πρέπει να τις στηρίξουμε για να αναπτύξουν ανταγωνιστικές ε, προτάσεις και αιτήσει και όταν μιλάμε για αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους κοιόδες εισηγητές, ο κύριος Καντσιάν. Για την Επιτροπή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία λεπτά έχετε, λέει Πρόεδρος. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να εκφραστούμε σωστά. Πρώτον, γενικά θα ήθελα να πω ότι η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εγγύησης και με τα ομόλογα έργου και με τα ειδικά ταμεία σε μεμονωμένους τομείς. Ακόμα και αν δεν φτάσουμε στο ανώτατο όριο που επιθυμούμε, θα πρέπει να έχουμε εγγυήσεις για τη χρήση αυτών των μέσων και δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε εκ των προτέρων την εφαρμογή του. Εγώ πιστεύω στα μέσα αυτά γιατί φέρνουν σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα κάνουν τον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει και εκτός από το, το θέμα της μόχλευσης ε, υπάρχει ε, αποτέλεσμα. Για το θέμα της ενέργειας συμφωνώ με την εισηγήτρια. Νομίζω ότι ο προπολογισμό για την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες θα πρέπει να παραμείνει και να χρησιμοποιηθεί με τον πιο χρήσιμο τρόπο προωθώντας κυρίως τα καινοτόμα όπως είπα χρηματοδοτικά μέσα. Γι' αυτό η πρόταση για τον προϋπολογισμό είναι πολύ σημαντική να δούμε τι χρήματα θα υπάρξουν. Για την ενέργεια νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε τους καινοτόμους ε, τρόπους παραγωγής ενέργειας. Για τις μεταφορές άκουσα την εισηγητή. Έχω ήδη θέσει το θέμα των λεωφόρων της θάλασσας θα πρέπει να βρούμε τρόπο έτσι ώστε να ευνοήσουμε και τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα με άλλα μέσα. Αυτό θα διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές. Δεν μπορούμε να τις βοηθήσουμε αν δεν ε, λάβουμε σωστά υπόψη και τον συμβαλόμενο τώρα για τους διαδρόμους. Δεν βλέπω τι γίνεται σε επίπεδο διακυβέρνησης. Δεν μιλάμε για ένα τρίτο επίπεδο ε, προγραμματισμού. Πρέπει να βρούμε ε, σωστή διακυβέρνηση, πρέπει να διευκρινίσουμε τους διαχειριστές ε, συντονιστές αυτών των δικτύων. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τα τοπικά προβλήματα και θέματα και να προωθήσουμε την ιδέα των διαδρόμων. Τα τελευταία χρόνια ακούσαμε τις απόψεις των συντονιστών οι οποίοι πραγματικά εκφράζουν θα έλεγα μια αδυναμία στον τρόπο λειτουργίας. Ε, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις λεπτομέρειες, τις τοπικές. Το σύστημα έχει σημασία. Το σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι απαραίτητη έτσι ώστε να υπάρξουν εγγυήσει για την ομοιογενή ανάπτυξη των οικονομικών πόρων. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της τελευταίας φάσης. Θα έλεγα ακριβώς σε αυτή τη φάση μπορούμε να καταστήσουμε κερδοφόρους όλους αυτούς τους διαδρόμους και να καταστήσουμε χρήσιμα τα βήματα που κάνουμε στη διαχείριση των ροών μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάθε βήμα έτσι ώστε να συνδέσουμε αυτούς τους κόμβους με τις ροές. Ευχαριστώ τον κύριο Καντσάν. Πάντα σεβόμενοι τα τρία λεπτά έχει ο κύριος Πυρίλο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι τροπολογίες πάνω στις οποίες θα ξεκινήσει μια μελέτη σε βάθος ε, είναι οι σχετικές ε, στο άρθρο 7 παράγραφο 3 για την επιλεξιμότητα προγραμμάτων κοινού συμφέροντος τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και λίγες εβδομάδες στην Επιτροπή Ήτρε ψηφίσαμε την έκθεση του συναδέλφου Κάμπος για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές υποδομές. Σε αυτή την έκθεση προσετέθηκε μια συμβιβαστική ε, λύση για το άρθρο 15 που καθορίζει τα κριτήρια σχετικά λοιπόν με την χρηματοδότηση αυτών των κοινού ε, ενδιαφέροντος προγραμμάτων. Δεν θα σχολιάσω πολύ την συνένεση στην οποία καταλήξουμε χρηματοδοτούμε προγράμματα και πέραν του CCS, αλλά νομίζω ότι κάποιες αποφάσεις αυτές δεν είναι πολύ σωστές για δύο λόγους. Πρώτον, διότι διαψεύδουν ουσιαστικά αυτό το οποίο εμείς έχουμε εγκρίνει στα πλαίσια της Ήτρε μέχρι τώρα και δεύτερον εξασθενούν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο υπερψηφίζοντας τη συμβιβαστική αυτή πρόταση ε, έδωσε έντολη στους συναδέλφους για τον τριμερή διάλογο. Είναι δύσκολο να αποκατασταθούν οι συνέργειες στον τομέα αυτό. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε μια συμβιβαστική λύση για τη μείωση των ποσοστών συγχρηματοδότησης, όπως επίσης και την αύξηση κατά 10 ποσοστιαίων μονάδες των δράσεων που επηρεάζουν θετικά τον περιορισμό ε, των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών κτλ. Έχουν κατατεθεί επίσης και αρκετές τροπολογίες ε, για τους υπόλοιπους πόρους, για τον γεωργικό τομέα, ε, που εφόσον υπάρχουν υπόλοιπα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στους τομείς αυτούς. Έτσι θα μπορέσουμε να χρηματώσουμε περισσότερα προγράμματα. Θα υπάρξει μείωση και του πολιετούς ε, χρηματοοικονομικού πλαισίου, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος ορισμένων στρατηγικών προγραμμάτων. Μία επιπλέον παρατήρηση. για τις τηλεπικοινωνίες. Σε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί, οι τηλεπικοινωνίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μόνο από χρηματοδοτικά καθαρά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι στον τομέα αυτό θα δώσουμε την δυνατότητα να αποφασίσει πώς θα συλλέξει κάποιες επενδύσεις μόνο επί τη βάση του οικονομικού συμφέροντος, ενώ οι περιοχές της από από απομεμακρυσμένες περιοχές, οι ορεινές περιοχές δεν παρουσιάζονται σαν ιδιαίτερα ελκυστικές για επενδύσεις, διότι δεν είναι πυκνοκατοικημένες. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι και για αυτές τις περιοχές είναι απαραίτητες άμεσες επιδοτήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Πυρίλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει. Είναι πολλές τροπολογίες. Θα ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις. Έχουν κατατεθεί πάρα πολλές ε, ε τροπολογίες για τα παρατήματα και νόμιζα πως υπήρχε μια συμφωνία κυρίων για να μην κατατεθούν πάρα πολλές τα παραρτήματα, αλλά υπάρχουν ε, πάνω από 100 παραδείγματο χάρη για τους διάφορους διαδρόμους και αναρωτιέμαι πραγματικά ποια, πώς θα κριθεί το ποια είναι τα σημαντικά έργα για την ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερη παρατήρηση, οι τροπολογίες οι οποίες ε, εξασθενούν ε, την πρόταση της Κομισιόν ε, θα μου φανεί δύσκολο να την στηρίξουμε. Παραδείγματο χάρη η αρχή Use it or Lose It. Ίσως μου είναι πιο ενδιαφέρον αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν για κάποιο ανταγωνισμό, δηλαδή όποιος έρθει πρώτος θα εξυπηρετηθεί και πρώτος. Επίσης σημαντικό είναι να δούμε πραγματικά το ποστό χρηματοδότησης για να ληφθεί υπόψη και οι νέες τεχνολογίες ε, και η καινοτομία και να δημιουργηθεί βεβαίως να δημιουργηθούν και ίσοι όροι ανταγωνισμοί όσον αφορά τις ε, διάφορες ε, τεχνολογίες και τους, τα διάφορα μεταφορικά μέσα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε εισόδημα. Τέλος, για τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, η πρόταση της Κομισιόν ήταν νομίζω καλή και θα μπορέσουμε, ελπίζω, να βρούμε ε, μια συμβαστική λύση και θα πρέπει νομίζω να βρεθεί μια συμβαστική λύση η οποία θα είναι και ε, διαφανής ε, και σωστή και να μην αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών διαξυφισμών για να χαθούν αυτά τα 10 δισεκατομμύρια. Εν ολίγης νομίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε ε, ικανοποιητικούς συμβασμούς για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη γιατί είναι σημαντικά αυτά τα έργα, υπάρχει ευρωπαϊκή προσέμενη αξία, θα ωφεληθούν τα κράτη-μέλη και πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να στηρίζουμε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ τους ε, εισηγητές. Δεν είναι εύκολο με τόσο τροπολογίες να βρουν συμβαστικές ε, προτάσεις. Κοιτάξτε, ε, βλέπουμε πως έχουμε παραμείνει σε αυτά τα οποία θέλουμε. Ο καθένας έχει γράψει τις επιθυμίες του εδώ πέρα. Όλοι θέλουν να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πως δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση. Οπότε, εάν είχαμε ε, πει πως πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη συγχρηματοδότηση, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα πάρα πολλά έργα. Γιατί έχουμε και τα πολλά και τα μεγάλα. Να πω κάτι παραδείγματο χάρη για το τούνελ ε, στο, στη βάση του Μπρένερο. Κοιτάξτε, ε, είναι 65 χιλιόμετρα, από τα οποία πρέπει να σκαφτούν άλλα 35. Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν, είναι μηχανήματα. Και το εάν θα μετατοπιστεί η κίνηση έτσι από το δρόμο στο σιδηρόδρομο, είναι κάτι το αμφισβητούμενο. Εμεί θέλουμε χρηματοδότηση τη οικολογική αηφορία, θα δούμε πώ θα κερδίσουμε βέβαια και λεφτά εκ των υστέρων με τα έργα και πόσε δουλειέ θα δημιουργηθούν. Εάν είναι να υπάρξουν ε, βεβαίως οικοδομικά έργα. Γιατί τι θα χρησιμοποιηθούν τεράστια μηχανήματα ή θα χρησιμοποιηθούν άνθρωποι. Σημαντικό είναι επίσης να δούμε τα διασυνοριακά κομμάτια γιατί ξέρουμε πως δεν έχουμε ακόμα διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο και το κενό είναι ακριβώς στις μεθοριακές περιοχές και κανείς δεν βγάζει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Τα κενά που δημιουργήθηκαν και οι καταστράφηκαν στον πόλεμο και στη μεταπολεμική εποχή πρέπει εκεί να χρηματοδοτηθούν, γιατί δεν υπάρχει οπωσδήποτε εθνικό, το οποίο επίση δεν έχει μπει εδώ πέρα επί τη αρχή, γι' αυτό έχουμε κάνει και τι τροπολογίε μα. Η Αγιάλα Σέντερ είπε το θόρυβος δεν είναι τόσο θόρυβος. Μα εγώ θεωρώ πως εξοικονομούμε λεφτά με το να καταπολεμήσουμε το θόρυβο στην πηγή. Τα 10 δισεκατομμύρια ε, υπάρχουν εκεί πέρα για τι να σας πω για το Offenburg, που φτιάχνουν ένα τείχος για την καλομή στο Ρίβου 10 μέτρων, 10 μέτρων ύψους, δηλαδή ψηλότερο από το τείχος του Βερολίνου όταν υπήρχε. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι και στην καταπολέμηση του θορύβου στην πηγή. Κερδίζουμε σε τρεις ε, τρόπους εκεί πέρα, και χρόνο και χρήμα και είμαστε αποτελεσματικοί. Και βεβαίως Λίγα πράγματα, όπως είπα, ε, διαγράφηκαν. Εμείς διαγράψαμε κάποια πράγματα στα σιδηροδρομικά. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα από το κανάλι Ρήνου Μάιν Δούναβη. Το ακριβότερο τότε δημόσιο έργο της Γερμανίας που είχε πει ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων πως είναι το πιο ηλίθιο έργο που έχει γίνει από τον πύργο της Βαβέλ και Δόθε. Δεν είναι δυνατόν. Ε, και εδώ πέρα βλέπουμε εκατοντάδες εκατομμυρίων γιατί κοιτάξτε, βλέπει, πρέπει να το δούμε εμείς. Ε, εντάξει, 80% της εσωτερικής ναυσιπλοείας είναι στον ε, Ρήνο. Αλλά τώρα σύνδεση με τον Έλβα και τα λοιπά δεν είναι πάρα πολύ λογικά. Επίσης, είπα και οικολογικά και οικονομικά κριτήρια. Είπα, σας είπα λοιπόν, στα ε, μεθοριακά σημεία θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίσει να αναπτύσσεται μαζί και όχι να αυξάνονται τα κοινά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πόστελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαβάσω τη γνώμη του εισηγητή μας, του Σίλα. Ε, δεν είναι μαζί μας σήμερα, ζητεί γνώμη. Θέλει να ευχαριστήσει τους εισηγητές ε, και περιμένει να συζητηθούν τα θέματα αυτά τις επόμενες εβδομάδες. Καταρχήν θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την υποστήριξή μου στο μηχανισμό, στην διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, που δίνει πραγματικά προστιθέμενη αξία στις υποδομές ε, μεταφορών τηλεπικοινωνιών. Ε, και εσύ υποστηρίζει επίσης τις προτάσεις των συνσηγητών, ενώ υποβάλλει συγκεκριμένες τροπολογίες για βελτίωση της νομοδότησης. Σε ό,τι αφορά τους διαδρόμους, οι προτάσεις να δοθεί προτεραιότητα στους διαδρόμους θα πρέπει να, υποστηριχτεί, να υποστηριχτεί. Η ανάπτυξη των διαδρόμων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα έτσι ώστε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό του δικτύου. Σε ό,τι αφορά την ε, δέσμευση των 10 δισεκατομμυρίων των, του Ταμείου Συνοχής, ε, η δέσμευση αυτή θα πρέπει να παραμείνει και θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ε, η κατανομή ανακράτως μέλος θα πρέπει να σέβεται τις εθνικές οροφές αλλά ε, το σχετασία θα πρέπει να τα διαχειρίζεται κεντρικά η Κομισιόν. Ε, υπάρχει επίσης ένας βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των, ένας βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών θα βοηθούσε. Οπότε τα ποσά τα οποία δεν θα έχουν καταναλώσει τα κράτη-μέλη, απορροφή στα κράτη-μέλη μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση θα έπρεπε να διατεθούν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτό θα έδινε κίνητρο στα κράτη-μέλη να υποβάλουν προτάσεις. Τέλος, ε, θα πρέπει να καταστεί σαφές ε, ότι η κατανομή των κονδυλίων δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο 2,5% του ΑΕΠ σε οποιαδήποτε άλλη ε, οροφή ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο ένα ολόκληρο project θα μπορούσε να παραλύσει επειδή ο ένας ε, συμμετέχουν σε ένα κράτος μέλος έχει φτάσει στην οροφή του, στο νοτατόριο. Και δύο ακόμα σχόλια δικά μου. Ε, θεωρώ ότι ε, θα πρέπει οι επενδύσεις να γίνουν πολύ προσεκτικά στις ε, παρούσες τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες. Οι δαπάνες θα πρέπει οπωσδήποτε να εστιάζονται στην βιώσιμη ανάπτυξη ε, και ε, θα πρέπει να προσφέρουν ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης χαιρόμαστε που η Κομισιόν προσπαθεί να απλοποιήσει της, το σύστημα χρηματοδότησης. Δεν είμαι σίγουρη όμως ότι ε, η, ο κανονισμός η, ταυτόχρονη ε, εφαρμογή του, ε, μηχανισμού αυτού και του κανονισμού των ταμείων συνοχής θα βοηθήσει. Επίσης είναι σημαντικό ε, να ενταχθούν και τα χρηματοδοτικά μέσα έτσι ώστε να μειωθεί ο προπολογισμό, όχι να αυξηθεί. Ε, τέλος, η κατεξουδότηση ε, πράξεις δεν θα πρέπει να είναι τόσο πολλές, θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο λόγος των Κλωτ Τούρμες. Ε, θα είμαι σύντομος και θα προσπαθήσω να εστιάσω σε συγκεκριμένα σημεία ε, Η πρόταση του Συμβουλίου για τον Περιπολογισμό την περασμένη εβδομάδα μπορώ να πω ότι είναι προσβολή. Και το λέω με μετριοπαθώς ή ο προπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία ε, και ακριβώς είναι αυτό που κάνει. Ε, παρόλο που είναι αυτό το οποίο μας κατηγορούν δεν κάνει. Ε, είναι όλα τα προγράμματα που έχουμε προβλέψει είναι ευρωπαϊκά προγράμματα ευρωπαϊκής προστέμενης αξίας. Όλα αυτά μας τα κόβουν. Ενώ δεν κόβουν την γεωρική πολιτική, τα διευθυντικά ταμεία κλπ. Γιατί, γιατί προφανώς έχουν σχέση με την ε, με τις άμεσες εθνικές δαπάνες ε, και την επικουρικότητα. Θα πρέπει να πολεμήσουμε ενωμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ε, το ποσό το οποίο είχαμε χωρίς περικοπή, χωρίς την περικοπή αυτού του 40%, 40% είναι πραγματικά μια προσβολή. καταστρέφουν την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Δεν την υποστηρίζουμε αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Χρειάζονται υποδομές ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για υποδομές φυσικού αερίου. Γιατί έχουμε μια οδηγία ασφάλειας ε, εφοδιασμού φυσικού αερίου που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε υποδομές φυσικού αερίου. Αυτό έχει γίνει. Έχουμε βελτιστοποιήσει το δυναμικό μεταφοράς ε, των ε, υπαρχόντων ε, αγωγών φυσικού αερίου και δεν πιστεύω ότι η ζήτηση φυσικού αερίου θα αυξηθεί δραματικά τα επόμενα χρόνια. Βρισκόμαστε στο μέγιστο αυτή τη στιγμή γιατί η μεγαλύτερη χρήση φυσικού αερίου που γίνεται στα κτίρια θα μειωθεί. Θα μειωθεί αυτή η ζήτηση διότι ανακαινίζουμε τα κτίρια με τρόπο πιο οικολογικό, συνεπώς θα δαπανούν λιγότερο φυσικό αέριο, συνεπώς δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά χρήματα για το φυσικό αέριο. Τα, το μεγαλύτερο ποσό θα πρέπει να πάει στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερον, οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είναι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Ε, έχουμε ένα επενδυτή, ε, θέλει να επενδύσει για 50 χρόνια, οπότε αυτό ε, διαπραγματεύεται με τον ρυθμιστή, με την αρχή ρύθμισης, την τιμή. Ε, η χρηματοδότηση θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό και μόνο για πολιτικά συσσαγωγικά project. Για παράδειγμα, οι βαλτικές χώρες να γίνουν ανεξάρτητες ή λιγότερο εξαρτημένες από τη Ρωσία. Έχει πολιτική σημασία, ποτέ δεν πρόκειται να είναι οικονομικά βιώσιμο, εμπορικά βιώσιμο ένα τέτοιο project. Δεν μπορούν να γίνουν τόσο πολλές επενδύσεις. Εκεί ναι, να ε, ε, χρηματοδοτήσουμε, να επιδοτήσουμε ε, αλλά ε, να περιοριστούμε σε τέτοιου είδους πολιτική ή ζητήματα. Και τέτοιου είδου ε, project θα πρέπει να αποτελέσουν παράγοντες μόχλευσης για να ε, συγκεντρωθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Έχω επίση υποβάλει τροπολογίες για το εξή. Έχουμε ένα θέμα ε, κινδύνου κεφαλαίου. Στην Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία ε, τα επιτόκια είναι πάρα πολύ ψηλά, ενώ σε άλλες αγορές είναι πολύ πιο χαμηλά. Και χρειάζεται να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή οι αγορές ε, ε, επιβαρύνουν συγκεκριμένες χώρες. Και αυτές οι χώρες θα μείνουν πολύ πίσω, γιατί είναι πολύ ακριβό να ανανεωθεί, να ανακαινιστεί ε, η υπάρχουσα υποδομή, να εξυγχρονιστεί η ενεργειακή υποδομή. Συνεπώς πρέπει να βρούμε ένα, μια λύση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Allora adesso noi abbiamo ancora 13 interventi. Eh, Έχουμε 13 ακόμα ομιλητές στον κατάλογο. Εδώ κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Trautmann, Grandes, Liberazzaski, Vidal Quadras, Ertug, Vandalen, Prodi, Ticau, Galler, Correra do Campos, Caumazzalos. 14. Ancora? Ecco, 15. Per cui se vogliamo... 15 τελικά. Αν θέλουμε ε, να δώσουμε το χρόνο στους για να απαντήσουν, παρακαλώ να περιοριστούμε στο 1,5 λεπτό. Πολύ αυστηρά όμως. 1,5 λεπτό. Κύριε Τελκαστήγιο. 1,5 λεπτό λοιπόν. Πρώτον, υπάρχει ένα πρόβλημα με την έκθεση. Ε, δεν έγινε απαρκή συντονισμό τη συζήτηση. Συνήθω συζητούμε την έκθεση πλαίσιο και μετά τις ειδικέ εκθέσεις. Δεν είναι δυνατόν οι ειδικέ εκθέσεις και ιδιαίτερα σε αυτή τη ενέργεια και μετά των τηλεπικοινωνιών να ε, μπαίνουν στην διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο μέσω του τριμερούς διαλόγου και να μην έχουμε διαπραγματευτεί την, ε, το, την έκθεση που είναι ε, πλαίσιο. Η έκθεση αυτή έχει επηρεαστεί από αυτήν την κατάσταση. Να συγχαρώ τους συζητητές γιατί η η εργασία ήταν πολύ δύσκολη. Αυτό το σημείο το οποίο υπογράμμισα είναι σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνολικό προπολογισμό, θα πρέπει να είμαστε ε, ακαμπτοί και αν θέλουμε να γίνει κάποια μείωση, θα πρέπει να γίνει αναλογικά σε σχέση με αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Δηλαδή, αν μειωθεί το συνολικό ποσό, θα πρέπει αυτή η μείωση αναλογικά ε, να εφαρμοστεί σε όλα. Τέλος, την ενέργεια και τα ενεργειακά δίκτυα. Ψηφίσαμε και είναι υποδιαπραγμάτευση ε, το ότι τα προγράμματα θα ε, χρηματοδοτούνται είτε από επιδοτήσεις είτε από χρηματοδοτικά όργανα χωρίς πριοτεραιότητες και χωρίς ποσοστά. Το ίδιο θα ψηφίσουμε και σήμερα μετά από αυτήν εδώ τη συνάντηση σε ό,τι αφορά τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Σε αυτή την γραμμή θέλω να κινηθούμε, τουλάχιστον η δική μου ομάδα προς τα εκεί θα κινηθεί και για την έκθεση πλαίσιο. Ελ Καντράουι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και τους συζητητές για τη δουλειά που έκαναν. Κάποια πραγματάκια, βεβαίως πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εισηγητές όταν θα κρίνουν τις ε, τροπολογίες να εφαρμόσουν αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και για τα παραρτήματα γιατί θα πρέπει όπως είπα να χρησιμοποιήσουμε τα κονδυλιά μας στο μεγαλύτερο βαθμό για έργα με ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Επίσης να δούμε τα της συνοχής και όσον αφορά τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Αλλά σημαντικότερο είναι βεβαίως το πολιτικό μήνυμα όπως ε, το έχει ε, δώσει η Κυπριακή Προεδρία στον αφορά τον προϋπολογισμό και βεβαίως οι συνάδελφοι άσκησαν ε, κριτική γιατί είναι πάρα πολύ ωραία να λέμε πως θέλουμε στρατηγική ή να φροντίσουμε τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας και να μην υπάρχουν μετά στο τέλος κονδυλία. Πρέπει λοιπόν ε, να ορίσουμε τις προτεραιότητες μας, αλλά εγώ θα ζητούσα από την Κομισιόν όταν, εάν ε, το τελικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό το οποίο προτείνουμε, να μας πει η Κομισιόν ειλικρινά ποιες προτάσεις πρέπει να διαγραφούν. Γιατί πρέπει να πούμε ειλικρινά στον ε, πολίτη στην Ευρώπη που μπορεί και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη επενδύσεις τα επόμενα χρόνια και να προτείνει μια στρατηγική προς το Συμβούλιο για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο με αυτά τα λεφτά. Σας ευχαριστώ. Γκρος, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτά τα οποία είπαν. Σύντομα τώρα για την πρόταση της Προεδρίας του Συμβουλίου. Νομίζω πως είναι απλό. Το μοναδικό μέσο όπου υπάρχει ανάπτυξη και προσπαθούμε να επιτύχουμε τη στρατηγική του 2020 ε, είναι αυτό το οποίο περικόπτεται. Ε, αυτό είναι αναξιοπιστία. Εάν αυτέ οι αποφάσει που λαμβάνει το Συμβούλιο δεν είναι σωστέ. Επίση και το μοναδικό μέσο το οποίο αυτή τη στιγμή ε, επίσης ε, είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένα έργα είναι αυτό το, το ΣΕΦ. Και ο κάθε υπουργό, είτε είναι υπουργό μεταφορών είτε οτιδήποτε, μπορεί να πάει στη χώρα του και να πει Αυτό επέτυχα εγώ για τη χώρα μου, αυτά τα έργα εδώ πέρα τα μέσα, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα είναι πράγματι σημαντικά, αλλά και παίζει και το εξή ένα ρόλο. Εάν θέλουμε να έχουμε επενδυτέ πλην του δημοσίου, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι και πιστικά τα έργα τα οποία προτείνουμε και να μην υπάρχουν και αυτές οι αμφιβολίες γιατί αυτό το μέσο το οποίο έχουμε μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης το Ταμείο Συνοχής Νομίζω πως ε, είναι σε καλό δρόμο. Χρειαζόμαστε αυτό το συμβασμό μεταξύ της Επιτροπής ε, Ρέγγι και της δικής μας, ότι δηλαδή θα εργαστούμε με φακέλους, θα έχουμε την αρχή use it or lose it, γιατί πρέπει να υπάρξει μία πίεση και βεβαίως θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε να γίνει μία αρχή με τους νέους φακέλους. Τώρα, για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και όλες αυτές τις όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Έχουμε μια γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπήρχε μια συνένεση μεταξύ Κοινοβουλίου, Χωρών και Κομισιών, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε και προς τα έξω. Σας ευχαριστώ, Τροτμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ζητήματα βασικά. Το πρώτο έχει ήδη υπογραμμιστεί από πολλούς ομιλητές σε ό,τι αφορά το συνδυασμό των τύπων χρηματοδότησης ε, με ανησυχή η τροπολογία 59 που θέλει να ε, διαγραφεί η δυνατότητα χρηματοδότησης με δύο τρόπους ε, από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Φέρμ ζήτησε να διατηρηθεί αυτός ο διπλός τρόπος χρηματοδότησης. Δεύτερον, τροπολογία 47 που αναφέρει ότι η χρηματοδότηση ε, των δικτύων, ε, βριζονικών δικτύων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα. Είναι περιοριστικό. Ε, περισσότερο από τον τομέα της ενέργειας, οι επενδυτές εδώ πέρα είναι πιο διστακτικοί. Και δεύτερον, αν για τις περιοχές που καλύπτονται λιγότερο και που αναφέρονται στην έκθεση του κοινόβουλίου μας που είναι ε, περιοχές προτεραιότητας. Αν δεν μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και με επιδοτήσεις θα δυσκολευτούμε. Τέλος, ε, μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, που έχει στα χέρια της τα χρηματοδοτικά μέσα. Θα ήθελα να ακούσουμε την άποψή της για το ποιος θα είναι ο ρόλος της με βάση τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ. Ο λόγος του Τεγκράντης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα περιοριστώ στα θέματα των μεταφορών. Γιατί υπάρχουν ειδικοί για τα υπόλοιπα. Καταρχήν συμφωνώ με την κριτική που εκφράστηκε σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας για τον προπολογισμό. Και πάλι έχουμε ε, μια χαμένη ευκαιρία με αυτά τα νούμερα δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας, δεν υπάρχει περίπτωση να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίδεται. Τρίτον, θέλω να συγχαρώ τους συζητητές. Επέδειξαν λογική, σοφροσύνη, συνεπώς τους αξίζουν τα συγχαρητήρια. Τρία θέματα θέλω να τονίσω. Καταρχήν, η διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ήδη αναφέρεται στην έκθεση. Θα ήθελα όμως να αναφερθούμε και στα σύνορα των κρατών μέλων. Ε, δεύτερον, η σύνδεση με τους σιδηροδρομικούς διαδρόμους. Έχουμε συμπεριλάβει ε, την, την διαδρομή μέσα από τα Πυρηναία που συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό δίκτυο. Υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, δεν είναι δυνατόν να χάσουμε συγκεκριμένη χρηματοδότηση που ήδη υπάρχει. Ε, και τέλος, η αναθεώρηση των παρατημάτων θα γίνεται μαζί με, τα κράτη-μέλη. Δεν συμφωνούμε να γίνεται με κατεξουδότηση πράξη όπως προτείνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λόγω του κύριο Ριμπεράτσκι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Αγία Λασάντερα αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές. Πρέπει να θυμόμαστε πως το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη είναι μια κοινοτική μέθοδος. Αν προσθέσουμε και το Ταμείο Συνοχής, μιλάμε πως ε, έχουμε για μια διπλή προσταμινή αξία, δηλαδή τους διαδρόμους και την ε, συνοχή. Προσφάτως ε, ήμασταν υπέρ της επαναβιομηχάνησης της Ευρώπης, οπότε είμαστε οπωσδήποτε υπέρ των σιδηροδρόμων, των λιμανιών κτλ. Τώρα, αν μειώσουμε το συνολικό ποσό το οποίο θα πήγαινε σε αυτά τα έργα, αυτό σημαίνει πως χάνουμε την ε, αξιοπιστία μας, πως ε, λέμε αφενός δηλαδή πόσο σημαντική είναι η βιομηχανοποίηση και μετά ε, η βιομηχάνηση για την άλλη δεν δίνουμε λεφτά. Αν είναι λοιπόν να είμαστε σοβαροί, όπως είπε και ο κύριος Φέρμ, εμείς θεωρούμε πως σε αυτή τη φάση πρέπει να φροντίσουμε κάποια κονδύλια να παραμείνουν όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βιντάλ Κουάντρας. Θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα για την ενέργεια όλα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την ορολογία μιλάμε για τον μηχανισμό σύνδεσης διασύνδεσης Ευρώπης. Δηλαδή κατασκευή ε, υποδομών που, έχουν, που αποσκοπούν στην ενοποίηση της ε, Ευρώπης. Υπάρχουν και άλλοι ε, στόχοι της ε, πολι, ε, πολιτικής. για παράδειγμα, μείωση των εκπομπών, πρόθεση των ανανεώσιμων, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη βελτίωση των υποδομών. Και παρακαλώ να το θυμόμαστε. Δεύτερον, είναι ζωτική σημασία να ε, σταματήσουμε πλέον να ε, διαθέτουμε, να έχουμε ενεργειακά νησιά που να μην συνδέονται με τον υπόλοιπο κορμό της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά δίκτυα. Είναι σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των, των σχεδίων. Και αν θέλουμε να καταργήσουμε ε, τα σημεία συμφόρηση ε, στις μεταφορές, σίγουρα το ίδιο πρέπει να γίνει και στην ενέργεια. Συνεπώς, ο ορισμός του σημείου συμφόρησης δεν θα πρέπει να είναι περιορισμένο στις μεταφορές, αλλά να διευρυνθεί και στον τομέα της ενέργειας. Και τέλος, θέλω να σχολιάσω τη σχέση ανάμεσα στον κανονισμό για τον οποίο ήταν εισηγητής ο κ. Κορέα Δεκάμπος και σε αυτόν τον οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή. Ε, τότε στον κανονισμό τον πρώτο, ε, συζητούσαμε για τα κριτήρια να θεωρηθεί ένα σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος. Τώρα μιλούμε για τους, για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Μην ε, ε, ξεχνάμε τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Αν θεωρούμε ότι κάναμε καλή δουλειά στον κανονισμό τον οποίο ήταν συγητής ο κ. Κορέδε Κάμπος, ε, μην αρχίσουμε τώρα να αλλάζουμε τη θέση μας για εκείνον. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση χωρίς όμως να χάνουμε από τον ορίζοντα αυτά τα οποία είχαμε πει στην προηγούμενη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σερτούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι να συγχαρώ τους συναδέλφους για το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη γιατί τονίστηκαν σημαντικά θέματα όπως παραδείγματο χάρη η σύνδεση με τη Λευκή Βίβλα των Συγκοινωνιών και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, επίσης η προώθηση των νέων τεχνολογιών, πάρα πολύ σημαντικό και επίσης αναφέρθηκε το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η εμπλοκή τους στα έργα. Αυτό υπάρχει και στο δικό μας το έγγραφο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις κατευθυντήριες γραμμές. Και αυτό το οποίο επίσης θέλω να πω επίσης ε, ως θετικό σημείο είναι πως έχει αναφέρει τις λεωφόρους της θάλασσας ε, ως σημείο προτεραιότητας. Δύο ακόμα σημαντικά σημεία να αναφέρω, αναφέρθηκαν. Το ένα είναι το θέμα του θορύβου στους σιδηροδρόμους ε, συνάδελφοι αναφέρθηκε πράγματι εδώ πέρα έχουμε μεγάλη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία γιατί πρέπει να σκεφτούμε τι όφελος έχουμε το να λέμε πως ε, θέλουμε να κάνουμε μεγάλα έργα και μετά σε εθνικό επίπεδο να μην μπορούμε να τα κάνουμε γιατί ε, υπάρχει ξέρω εγώ απαγόρευση κυκλοφορία στη νύχτα λόγω του θορύβου. Οπότε ειδικά στον τομέα του θορύβου πρέπει να υπάρξει μια συνοχή μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και της υφιστάμενης ε, νομοθεσίας και θέλω οι δύο εισηγητέ, οι συγκήτριες εδώ πέρα να το ξαναδούν το θέμα. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό και τελειώνω η εσωτερική ναυσιπλοεία και εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε βάρος και ολοκληρώνω ελπίζω να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε αυτά και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Συμβουλίου, αλλά βλέπω πως εδώ πέρα πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές... Ε, παρά το ότι είμαστε πράγματι κατά τη ε, τοποθέτηση του Συμβουλίου, έχουμε καταθέσει πάρα πολλέ ε, τροπολογίε στα παρατήματα. Οπότε πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το τι κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Κατόπιν, κυρία Πρόεδρε, με έκπληξη ε, πληροφορήθηκα τον, το πώς οι πράσινοι Γερμανοί και ο κύριος Κράμερ εδώ πέρα τοποθετήθηκαν όσον αφορά το μέλλον της εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας. Ο Δούναβης εδώ πέρα είναι ο κατεξοχήν ευρωπαϊκός ε, ποταμός, αλλά έχουμε καταθέσει κάποιες ε, έχουν καταθεθεί εδώ πέρα κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες αντικαθιστούν το Άμστερνταμ με, με την Αμβέρσα. Ε, τι να σας πω. Αυτά, εμείς θα τις ξαναδούμε αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρόντι. Συμφωνώ με τους καταλόγους για τις χερσές και τι ιδεονομικές μεταφορέ και για τι ενέργειες με κάποιε με ελάχιστε μικρέ αλλαγέ. Οι κανονισμοί για το, τις ενέργειες μεταφορές ε, ε, αναφέρονται στο ΣΕΖΑΡ ε, και θα πρέπει να προσθέσουμε επίσης και την, κυβερνο, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τους δορυφόρους θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε μέσα σε κρίση. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αυτές οι επενδύσεις να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε ε, στεναρά υπέρ της στήριξης των υποχρεώσεών μας. Και όταν ολοκληρωθούν οι υποδομές θα μπορούσαν ενδεχομένω και να ιδιωτικοποιηθούν. Ε, έρχομαι από την Κίνα, ε, επέστρεψα από την Κίνα πριν από λίγο και με εντυπωσίασε εκεί η, ε, το μέγεθος των επενδύσεων που γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η υλοποίηση, η εκτέλεση των έργων γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας και να προσαρμοστούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Τιτσάου, η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ε, μεταφορών και βέβαια από τις τεχνολογίες πληροφορίας. Συνεπώς δεν είναι αποδεκτό να μειώσουμε τον προπολογισμό δεν θα μπορούσαμε αλλιώ να υλοποιήσουμε την ψηφιακή ατζέντα. Θα πρέπει σίγουρα ε, να εξισωθεί η ανάπτυξη των δικτύων σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποδομές μεταφορών. Σε ό,τι αφορά την χρήση των 10 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Συνοχής, αυτό το ποσό, αυτό το κονδύλι θα πρέπει να δοθεί ε, με βάση τα εθνικά σχέδια και κατά αναλογία με αυτά. Οι επιδοτήσεις όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη και την γεωγραφική ποικιλία, όχι μόνο ε, θεματικά κριτήρια. Θα πρέπει επίσης το κανάλι μεταξύ του Μάιν και του Δούναβη να υποστηριχτεί σε ό,τι αφορά τα προγράμματα. Ε, επίσης η σύνδεση Μπρέιλα Ματσίν ε, που θα πρέπει να γίνει ε, ε, ε κόμβος μεταξύ ε, χερσαίων μεταφορών και σιδηροδρομικών μεταφορών ταχείας ε, ε, με υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Βουκουρεστή και Κωνσταντσα. Είναι πολύ σημαντικό για να καλυφθεί και η Μαύρη Θάλασσα που έχει ξεχαστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι ήδη κάποιοι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στο θέμα του θορύβου γιατί θεωρώ πως όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία πρέπει να δούμε και το να αποδέχονται οι πολίτες την πολιτική μας Γι' αυτό έχω μια συγκεκριμένη παράκληση προς την ε, εισηγήτρια, το θέμα αυτό του θορύβου να μην το δει έτσι δευτερευόντως, αλλά να διατηρήσει την δυνατότητα που πρότεινε η Κομισιόν να υπάρχει η δυνατότητα συγχρηματοδότησης για την προσαρμογή του τροχαίου υλικού για τη μείωση του θορύβου των σιδηροδρόμων γιατί το τροχαίο υλικό είναι αυτό το οποίο προκαλεί κυρίως τον θόρυβο και όπως είπα έτσι θα αυξηθεί η αποδοχή των ε, έργων μας γιατί όποιος έχει προσπαθήσει να διανυκτερεύσει δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή ξέρει πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχει απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας και αν είναι να πάει περισσότερη κυκλοφορία να μετατοπιστεί στους σιδηροδρόμους πρέπει να καταπολεμήσουμε το θόρυβο στην πηγή γι' αυτό σας παρακαλώ να μην διαγραφεί αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ. Ο Κορέιρα Ευχαριστώ πρόεδρε. Τέσσερα σημεία. Πρώτον, να ευχαριστήσω τους ηγητές για την δεκτικότητα που έχουν δείξει ε, για την ευελιξία τους. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε νομοθετικά συνεπείς, το είπε και ο Αλέχο Βιδάλ Κουάδρας. Δεν είναι δυνατόν το ένα στο ένα νομοθετικό κείμενο να χρησιμοποιούμε κάποια κριτήρια και σε ένα άλλο νομοθετικό κείμενο κάποια άλλα. Για παράδειγμα, άρθρο 15. Ε, ξαφνικά βγαίνει μια καινούρια προτεραιότητα με τον κανόνα του first coming, first First come, first serve, δηλαδή όποιο πρόγραμμα φτάσει εξυπηρετείται πρώτο. Ε, τρίτον, ε, για τη χρηματοδότηση έχω και εγώ μια τροπολογία, αλλά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα ε, να δεχτώ τη χρηματοδότηση της κυρίας Δελκαστήγιο για να μην αναφέρουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τέλος, αν γίνουν περικοπές, θα πρέπει να είναι αναλογικές. Αλλά ακόμα δεν έχουμε χάσει τον αγώνα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για υψηλότερα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κ. Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι δύσκολο, αλλά εγώ είμαι ένας εύκολος άνθρωπος όπως θα καταλάβετε από τις παρεμβάσεις που θα κάνω. Ε, Πέντε σημεία, πολύ γρήγορα. Πρώτον, υποστηρίζουμε όλοι τον χρηματοδοτικό μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη. Έχει τη στήριξη όλων μα και αυτό θα είναι ένα βασικό στοιχείο τη ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει μέχρι και την ψήφιση. Δεύτερον, η πρόταση ενό δραματικά περιορισμένου προπολογισμού, όπω αυτό που έχει κατατεθεί, αυτή η πρόταση που έχει κατατεθεί, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τόσο περιορισμένο προπολογισμό βάζει ουσιαστικά δυναμίτη στα θεμέλια της προσπάθειας που κάνουμε στα, δίκτυα, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ε, ενέργειας και επικοινωνιών. Δεν μπορούμε, αν δεν μπορούμε να διασώσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστήριξη στην ανάπτυξη, τουλάχιστον το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασώσει την αξιοπρέπειά του. Εάν κοπούν χρήματα από τον προπολογισμό, θα πρέπει αναλόγως να κοπούν και τα έργα που προβλέπονται. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο αλλά όπως υπόθηκε μόλις πριν από τον προλαλήσαντα συνάδελφο, ο αγώνας δεν έχει χαθεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τον δίνουμε με πίστη και επιμονή για να μην χάσουμε τα χρήματα τα οποία χρειάζεται, χρειάζεται μέσο των μεταφορών και γενικότερα η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τρίτο σημείο, στα επιμέρους ζητήματα. Υποστηρίζω την ενίσχυση της ανάπτυξης των διαδρόμων της θάλασσας, των motorways of the sea και αυτό, όπως και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε προτείνει την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από 20% σε 30%. Τελευταίο σημείο, κυρία Πρόεδρε. Τα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής. Ο μηχανισμός συνδέοντας στην Ευρώπη δεν μπορεί να τα στερηθεί αυτά τα χρήματα, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις των κρατών συνοχής. Οι, δύο συνάδελφοι, ο κύριος Δρικέ και η κυρία Γιάλα Σέντερ, πρέπει να βρουν έναν, έναν ένα συμβιβασμό που θα γίνει δεκτός από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει στο θέμα αυτό και έχω δύο σχόλια. Το πρώτο αφορά το θέμα Ταμείου Συνοχής. Ε, πρέπει να βρεθεί εδώ πέρα ένας καλός συμβιβασμός. Ε, είτε ε, διατηρώντας ε, τους εθνικούς ε, φακέλους είτε μέσω της διαφάνειας στην επιλογή ποιοτικών έργων που δεν χρειάζεται να βασίζονται στον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών. Το πρώτον αυτό και δεύτερον, συμφωνώ με αυτούς που είπαν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα των επιχορηγήσεων γιατί δεν μπορούν να υποκατασταθούν πλήρως από άλλα μέσα. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της εδώ με τρεις εκπροσώπους. Βέβαια δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Ακόμα και λιγότερο για να ακούσουμε και άλλους συγητές μετά. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει από σας. Εγώ θα αναφερθώ στο οριζόντιο τμήμα και στο τμήμα των μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω λίγο περισσότερο γιατί καλύπτω τα περισσότερα θέματα από αυτά που σας απασχολούν σήμερα, το Συνδέοντα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για την στήριξή τους, ιδιαίτερα στα πλαίσια και τη συνεισφορά της Κυπριακής Προεδρίας στη συζήτηση. Είναι σαφές ότι εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το τελευταίο κομμάτι του διαπραγματευτικού κοιτίου, όπως λέγεται, του negotiating box, για λόγους δημοσιονομικούς. Επίσης αυτό εμπλέκεται και με την αυξανόμενη κινητοποίηση των εμπλεκομένων στο μέσο αυτό. Υπάρχουν τουλάχιστον 600 που έχουν υπογράψει μία δήλωση, ανάμεσα σε αυτούς είναι και μέλη της Επιτροπής σας, αλλά και υπεύθυνοι επιχειρήσεων που θέλουν να παραμείνει το θέμα αυτό σαν ένα κομβικό για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της Ευρώπης. Τώρα ορισμένα οριζόντια σχόλια τηλεγραφικά. Οι τροπολογίες που τίνουν σε συνέργειες είναι θετικές, αλλά βέβαια μπορεί να υπάρξουν εκεί όπου έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές κατά τομέα και αυτό ισχύει για την ενέργεια για να είναι επιλέξιμη επίσης και η αγορά γεών. Αυτό έχει περιορισμένη θα έλεγα εμβέλεια και το ίδιο περιορισμένη είναι και η έννοια στη συγκεκριμένη περίπτωση της ε, μόχλευσης. Θα επανέλθω στα θέματα των μεταφορών. Ενθαρρύνουμε τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές να συμφωνήσουν στην μεταφορά των πιστώσεων από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μια χρονική διάρκεια συγκεκριμένη για τις χώρες συνοχής και θα επιτρέψει τον χρόνο να μεγαλώσει ο χρόνος ε, καταβολής αιτήσεων από πλευράς επιχειρήσεων και εμπλεκομένων γενικότερα. Απαιτείται να κρατήσουμε ένα σεφ το οποίο να είναι ε, θα έλεγα ευθυγραμμισμένο με τον προϋπολογισμό. Δεν θα πρέπει να μιλάμε σε επίπεδο διαπραγμάτευσης με ένα μειωμένο προϋπολογισμό. Θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουν οι συζητήσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο περιορισμός είναι δεδομένο στον προϋπολογισμό και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε στους στόχους που έχουμε. Πολλές από τις τροπολογίες λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά ταυτόχρονα ε, διευρύνουν το επίπεδο επιλεξιμότητας, αυξάνουν τα ποσά τα οποία θα ήταν θεωρητικά διαθέσιμα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θα εξασθενήσει την πολύ, ε, αν θέλετε, σωστά συγκεντρωμένη αρχική πρόταση. Κάποια επιπλέον συγκεκριμένα θέματα εμένουμε στο λεγόμενο κομβικό ή βασικό δίκτυο, το Core Network. Κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί το συνδέουν ε, αυτό το δίκτυο με διαμεθοριακές συνεργασίες, με επιμέρους εξελίξεις, με προηγούμενα κατά προτεραιότητα προγράμματα. Οι τροπολογίες αυτές είναι πολύ στοχευμένες, πολύ εξειδικευμένες, χρήσιμες τελικά. Αλλά παρόλα αυτά, αφού δεν έχουμε τα χρήματα που θα θέλαμε, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο κομβικό δίκτυο. Το ίδιο ισχύει επίσης ε, και τον λεγόμενο καθορισμό των bottlenecks και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε κομβική στόχη. Τώρα για τους θορύβους και τους ε, εξοπλισμούς οι οποίοι φέρονται στα οχήματα παντός είδους. Ε, δεν Υπάρχει η δυνατότητα για την χρηματοδότηση τέτοιων μέσων τα οποία θα φέρονται ε, στα αεροσκάφη κτλ. Γιατί αυτό λειτουργεί σαν μοχλός για την επίτευξη άλλων στόχων Πάντως ε, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και του ε, τροχαίου υλικού και των ε, υλικών γενικότερα και των εξοπλισμών γενικότερα σε όλους τους τομείς αυτούς των μετακινήσεων. Άκουσα κάποιες ιδέες σχετικά με την χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Πολλά μπορεί να χρηματοδοτηθούν από τον ιδιωτικό τομέα, όχι όμως όλα και εδώ έρχεται η περίπτωση του Σεζάρ Σχετικά τώρα με τις τροπολογίες στο παράρτημα 1. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν κατεθεί. Τα περισσότερα μέλη λένε ότι πρέπει να στοχεύσουμε συγκεκριμένες αρχές. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κεντρικό δίκτυο και τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα στην περίοδο 2014-2020. Αυτά και αν θέλετε για περιττέρω θέματα σε επίπεδο διμερές μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αν έχετε κάποιες περιττέρω ερωτήσεις, τώρα να δώσω το λόγο συναδέλφος. Κοιτάξτε, να μην δείξουν το ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος α, στην ενέργεια και στις λεπικοινωνίες. Λοιπόν, ένα λεπτό ο καθένας από, τα υπόλοιπου από τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μην ξεχάτε ότι ψηφίζουμε στις 5.30. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα περιορίσω τις παρατηρήσεις μου σε δύο σημεία. Καταρχάς θεωρώ τον προσανατολισμό των προτάσεων τροπολόγησης στον τομέα του ICT θετικές. Συμφωνούμε με αρκετές από τις τροπολογίες αυτές ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την βελτίωση των υποδομών. Εκεί έχουμε τις περισσότερες θετικές επιπτώσεις και την προστιθέμενη αξία. Υπάρχει εδώ και συγκεκριμένο σημαντικός χώρος θα έλεγα για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε μια κάποια εμπειρία. Πιστεύουμε ότι και μέσω της διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων περισσότερες επενδύσεις σε ευρώ θα βοηθήσουν να πενταπλασιαστεί και περισσότερο ακόμα οι επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Το για τα ΣΕΦ προφανές ε, είναι ότι στις αεροκατοικημένες περιοχές κάτι τέτοιο δεν ε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για θέματα στα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις, για την υψηλή ταχύτητα. Ε, Προφανώς οι επενδύσεις του ΣΕΦ που θα φτάνουν τα 100 μεγαμπίτη ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως έρχεται σε σύγκρουση με την υπεδίωξη της τεχνολογικής ουδετερότητας σε σχέση με τα φάσματα συχνοτήτων τα οποία θα καλύψουμε. Αν βάλουμε το επίπεδο πάρα πολύ υψηλά, ίσως να μην υπάρξει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν θα είναι υπαρκώς εμπορικά ελκυστικά τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστούμε την Επιτροπή λοιπόν. Α, έχουμε και την ενέργεια λέει η Πρόεδρος. Λίγα δευτερόλεπτα για την ενέργεια. Ευχαριστώ. Για την ενέργεια δύο σημεία θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, νομική συνεκτικότητα ανάμεσα στο ΣΕΦ και τις τομεακές κατευθυντήριες γραμμές, όπως το είπε και ο κύριος Κορέρε Κάμπος. Αυτό σημαίνει ότι θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων και δεν θα ανοίξουμε ε, το κουτί της Πανδώρας ε, ε, και σε άλλες ανάγκες χρηματοδοτικές. Χρηματοδότηση και σχέση ανάμεσα σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης και επιδοτήσεις. Πρώτον, θα υπάρχουν προγράμματα τα οποία οικονομικά θα είναι πολύ ισχυρά και τα οποία θα καλύψει η αγορά χωρίς πρόβλημα. Δεύτερον, θα είναι προγράμματα τα οποία είναι βιώσιμα εμπορικά αλλά τα οποία θα έχουν κάποια προβλήματα στην κάλυψη μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης. Σε αυτό το τομέα τα χρηματοδοτικά μέσα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, 10 με 15% του ΣΕΦ θα πάει προς τα εκεί, η τρίτη κατηγορία. Είναι θετικές εξωτερικές συνεισφορές στην κοινωνία και τις γειτονικές χώρες. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία εμπορικά δεν είναι βιώσιμα, και εδώ τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα βοηθήσουν γιατί δεν υπάρχουν τράπεζες οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους αν θέλετε στόχους όπως η λήξη της απομόνωσης, η περιφερειακή καινοτομία, η κάλυψη μεγάλων αποστάσεων κτλ. Οπότε εδώ οι επιδοτήσεις θα είναι απαραίτητες, θα συμπληρώνουν τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο λεπτά. Έχει ξανά το λόγο η Αγιάλα Σεντέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, που όχι μόνο υπέβαλαν τροπολογίες αλλά συμμετείχαν και στην συζήτηση για να διευκρινίσουν τις προτεραιότητές τους ε, και τις ίδιες τους τις τροπολογίες ελέγχθη ότι πράγματι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει και είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που θα βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης. Δεύτερον, πιστεύω ότι για τα διάφορα θέματα τα οποία σχολιάστηκαν. Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Έχουμε σχόλια για, τα οποία, για ορισμένα θέματα τα οποία μπορούμε να ε, ρυθμίσουμε. Για παράδειγμα με την ε, ηχορύπανση. Ε, ίσως θα μπορούσαμε τελικά να πληρώσουμε το τροχείο υλικό των εταιρεών, μια και η, ε, η απόφαση για τα μέσα θα λαμβάνεται ε, ε, ε, με βάση και αυτά τα κριτήρια. Καταλαβαίνω βέβαια τα κριτήρια, τα, τα επιχειρήματα ορισμένων συναδέλφων, αλλά μην ξεχνάμε ότι ε, μιλούμε για υποδομές. Αν μιλήσουμε για ε, οτιδήποτε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να οι συνάδελφοι οι οποίοι επιζητούν την επιδότηση του τροχαίου υλικού να μιλήσουν με τους ε, υπουργού τους ε, έτσι ώστε να μας ε, δώσουν περισσότερα χρήματα από πλευρά Συμβουλίου. Αν είχαμε μεγαλύτερα κονδύλια τότε θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και το τροχαίο υλικό. Τέλος, συμφωνώ με, την, με το διάδρομο των, κεντρικό διάδρομο των πυρηναίων η υποστήριξη αυτή θα μας βοηθήσει ε, και άλλου είδους ε, project ε, που μπορούν να προσθεθούν γιατί είναι δικαιολογημένα. Σε ό,τι αφορά την κυρία Δικαστήγιο, προφανώς η ενέργεια δεν είναι το δικό μου ζήτημα, αλλά όλα είναι σχετιζόμενα βέβαια. όμως δεν είναι αλήθεια ότι γίνεται η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε εντολή να μην κλείσουμε καμία διαπραγμάτευση αν δεν τις κλείσουμε όλες μαζί γιατί αλλιώ προφανώ θα δημιουργούσαμε προβλήματα σε αυτό τον χρηματοδοτικό κανονισμό. Ελπίζω αυτές οι διαπραγματεύσει, οποιασδήποτε διαπραγματεύσει που γίνονται, να μην είναι επίσημες, να είναι ανεπίσημες. Κύριε Ρικέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων και για τις παρεμβάσεις τους και για τις τροπολογίες και τις σκέψεις τους. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή προκαλεί, αυτές οι εκθέσεις μάλλον προκαλούν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται από τις παρεμβάσεις. Δύο πράγματα να υπογραμμίσω. Πρώτον, εγώ δεν άκουσα κανένα από τους συναδέλφους να λέει κάτι διαφορετικό από το ότι δεν δέχεται την πρόταση του Συμβουλίου και ότι είναι προσβλητική η πρόταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ την γενικότερη κινητοποίηση εναντίον της προτάσεως του Συμβουλίου η οποία είναι αμφισβητήσιμη και απαράδεκτη. Θα πρέπει μάλιστα να δούμε και τις θέσεις αναχώρα και να δούμε τι λειτουργικές συνέπειες έχει κάτι τέτοιο και τι συνέπειες ε, ε, θα έχει και στους φορολογουμένους των χωρών αυτών. Ένα τελευταίο να παρατηρήσω ότι απαιτείται να υπάρξει συγκέντρωση. Συγκέντρωση σε ένα νομοθετικό μέσο απλό, κατανοητό, το οποίο να είναι γρήγορα εφαρμόσιμο και να καταστεί ταχύτατα λειτουργικό. Δεύτερον θα πρέπει να συγκεντρώσουμε επίσης ε, την προσοχή μας σε συγκεκριμένους στόχους και να πάψουμε να διευρύνουμε τους στόχους και τα πλαίσια μέσα στα οποία θέλουμε να λειτουργήσουμε. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και σε γεωγραφικό επίπεδο και σε θεματολογικό επίπεδο και να καλύψουμε κάποια κενά εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και τρίτον να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των σχεδίων αυτών. Εδώ θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβαστικές προτάσεις έτσι ώστε να καταστεί το πρόγραμμα αυτό πυκνό και λειτουργικό τάχιστα. Η συνάδελφος Βαλεάννα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούσαμε πολλές ε, πολύτιμες ιδέες και έχω την εντύπωση πως ε, όλοι πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση για να έχουμε μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να επιτύχουμε την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών σε όλους τους τομείς που μας απασχολούν, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου πως το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει και συνέπεια και με άλλες εκθέσεις και είμαι σίγουρος πως ε, ε, ο κύριος Κορέας Τεκάμπους και οι άλλοι συνάδελφοι θα το φροντίσουν. Επίσης για την ε, Κομισιόν είμαι σίγουρος πως δεν θα χρησιμοποιήσει την πίσω πορτέλα την κανονική οδό για την νομοθεσία της και το ίδιο θα κάνει και τώρα και η Κομισιόν πρέπει να είναι συνεπής και με τον εαυτό της γιατί όταν λέει πως οι ανάγκες για υποδομές ε, ενεργειακές είναι 200 δισεκατομμύρια και η χρηματοδότηση του μέσου συνδέοντα στην Ευρώπη είναι 9 δισεκατομμύρια το πολύ και αυτό πάει σε επιδοτήσει το 90%. Ποτέ δεν θα φτάσουμε τα 200 δι που λέει η Κομισιόν πώς ε, χρειαζόμαστε για το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριο Σίμψον, αν θέλει το λόγο. Sorry, first of all, thank you. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενήσατε σήμερα το απόγευμα για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Ελπίζουμε ότι θα σας φιλοξενήσουμε στις 27 Νοεμβρίου όπου θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Ε, ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθειά σας. Ε, να ευχαριστήσω, να πω μάλλον στα μέλη της Δική μου Επιτροπής ότι θα πρέπει να περάσουμε στην αίθουσα 3ε2 για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι της Ήτρε παρακαλώ να παραμείνουν στην αίθουσα γιατί θα ξεκινήσουμε αμέσως με τις ψηφοφορίες. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα αμέσως.